Άρχεται η συνεδρίαση. Θα ήθελα να κάνω ορισμένε ενακτήριε παρατηρήσει. Πριν από πέντε μέρε πήραμε τα λυπηρά νέα του θανάτου του Χιλ Ζακέ, ενό Γάλλου δημοσιογράφου που σκοτώθηκε στην πόλη Χόμ τη Συρία. Πέρσι, πάνω από 100 δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή του. στο καθήκον τους, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του καθήκον Καθήκοντός τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πάντα την ελευθερία έκφρασης και θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε αυτούς οι οποίοι εργάζονται για την αποκάλυψη της αλήθειας. Τουλάχιστον έξι άτομα επίσης έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά από το ατύχημα του Ιταλικού κρουαζιερόπλου. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι ένα ατύχημα το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί και ελπίζουμε ότι θα μάθουμε τα αντίστοιχα μαθήματα από αυτήν την ναυτική καταστροφή. Έχουμε επίσης λάβει και την είδηση του θανάτου του Μανουέλ Φράγα Ιριμπάρνε με τον θάνατό του η Ισπανία και η Ευρώπη χάνουν ένα μεγάλο πολιτικό άνδρα, ένα από τους κύριους αρχιτέκτονες της, δημοκρατικής, της σύγχρονης δημοκρατικής Ισπανίας. Ήταν ηγέτης και ιδρυτής του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας, του Παρτίδο Ποπουλάρ, που οι ηγέτες του είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Ο Μανουέλ Φράγνε, Φράγα Ιδιμπάρνε ήταν ο ίδιος στη δεκαετία του 1980 μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, θα ήθελα μέσω της ε, κόρης του, της κυρίας Κάρμεν Φράγα Εστέρες, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του μετελθόντος. Τέλος. Στις 18 Δεκεμβρίου ο Βάτσλαβ Χάβελ απέθανε. Ήταν πρόεδρος καταρχήν της Τσεχοσλοβακίας και μετά για δύο θητείες της Τσεχικής Δημοκρατίας. Η Ευρώπη και ο τσεχικός και σλοβακικός λαός έχασαν το σύμβολο της Βελούδινης Επανάστασης και το σύμβολο της επανένωσης Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ήταν ένας θαραλέος πολιτικός άνδρας, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2009 μίλησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον χειροκρότησαν όρθιοι όλοι οι βουλευτές. Αποτείουμε φόρο τιμή στη μνήμη του. Εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Πράγα στην κηδεία του Βάσλαβ Χάβελ. Και ήταν πράγματι μια μοναδική εκδήλωση μια τελετή που εξέφρασε και την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια συνένεση σεβασμού προς τον Βάτσλαβ Χάβελ, τον μεγάλο αυτό τσέχο πολιτικό. Θα ήθελα τώρα αγαπητοί συνάδελφοι να σας ζητήσω να σηκωθείτε για ενός, για, ε, για ενός λεπτού σιγή εις τιμή των δύο αυτών μεγάλων πολιτικών ανδρών. Thank you very much. Ε, Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές. Βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού μας